Ξεκινάμε με την κοινή θέση Συμβουλίου της Αιτιολογήσης ε, και την κοινή θέση του Συμβουλίου. Ο τίτλος θα δημοσιευτεί στα σημερινά πρακτικά. Οπότε από αύριο ξεκινάει η τρίμηνη προθεσμία του Κοινοβουλίου από τις 16 Ιανουαρίου 2009. Ανακοινώνω επίσης πως τα μέλη Μάρτο Καπάτο Κουμπίτσκα, Τόμας Μακτάνο και Χέλγα κατέθεσαν